Ερχόμαστε λοιπόν σε επεξηγήσει ψήφου για την έκθεση Κάρας. Το λόγο έχει ο κύριος Στρέσεκ καταρχάς. Κύριε Στρέσεκ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω μια επεξήγηση ψήφου για την έκθεση Κάρας, ποιότητα στατιστικών στοιχείων. Είναι εξαιρετική έκθεση από πολλές απόψεις, αλλά εγώ απέσχον γιατί δεν συμμερίζομαι την άποψη του εισηγητή ότι η Eurostat πρέπει να παίζει κυρίαρχο ρόλο. με ευνίδιους ελέγχους στις στατιστικές υπηρεσίες και να παρακολουθεί το και να ελέγχει το έργο τους έτσι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Στρέσεκ. Κύριος Χάνων έχει το λόγο. Χάνων! Συγγνώμη, αλλά δεν σας άκουγα με όλο αυτό το θόρυβο, κύριε Πρόεδρε. Ε, αποσπαστεί η προσοχή σας κύριε συνάδελφε. Λυπούμε, λυπούμε. Κύριε Πρόεδρε, κακό να μιλά κανείς για τα γεγονότα στην Ελλάδα ως τραγωδία, αλλά νομίζω ότι πραγματικά μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε ως τραγωδία από την κλασική σοφόκλειο έννοια. Είχαμε την ε, χρονιές του λεγόμενου boom ε, της ανάκαμψης, ε, τώρα έχουμε την έμεση όμως από υπερβολική διόρθωση της αγοράς. Η κάθαρση ωστόσο έχει γίνει τεχνητή, χωρίς να επιτρέψει μια φυσική διόρθωση της αγοράς, δηλαδή να να επανέλθει με το δικό της νόμισμα η Ελλάδα στις ευρωπαϊκές αγορές. Εμείς ε, προτείνουμε καλύτερη στατιστικά, καλύτερα στατιστικά στοιχεία, περισσότερους φόρους ε, και ε, τέλος πάντων άλλα μέτρα για την αναβολή του αναπόφευκτου ουσιαστικά και οι Έλληνες και ίσως και οι πολίτες άλλων χωρών της Μεσογείου έχουν να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον δύο χρόνια ύφεση, αλλά δημιουργούμε και εμείς ε, ε, δικαιολογούμε την ύπαρξή μας ουσιαστικά. Το θέμα είναι να εξασφαλίσουμε την απασχόληση των πολιτών. Ο κύριος Καμάλ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν δούμε την ποιότητα στατιστικών δεδομένων κάποιων κρατών μελών, φαινόταν ότι τα μαγείρευαν και δεν αντικατόπτριζαν την ε, οικονομία. Καταλαβαίνω την ανάγκη βελτίωσης των δεδομένων και την έκκληση για αυτή. Όλοι το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να είναι καλύτερα στατιστικά στοιχεία. Αλλά αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται προσχηματικά για την οικονομική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, ούτε προσχηματικά ώστε η Κομισιόν να έχει πρόσβαση στους εθνικούς προϋπολογισμούς ενός κράτους μέλους πριν υποβληθεί στο κοινοβούλιο, το Εθνικό Κοινοβούλιο αυτού του κράτους μέλους. Μην με την κρίση και τα λάθη που έγιναν στην κρίση ως δικαιολογία για περισσότερη ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, αλλά για να μάθουμε διδάγματα από την κρίση, να συλλέγουμε καλύτερα δεδομένα και να νοικοκυρέψουμε τα του οίκου μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Τώρα περνάμε στην έκθεση «Ο Λέχνιτσακ». Καταρχάς, δίνω το λόγο στον κύριο Κέλαμπ. Κέλαμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υποστήριξα την ε, έκθεση για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής θάλασσας και χαίρομαι που εγκρίθηκαν οι τροπολογίες μου. Πάντως σε συγκεκριμένα σημεία θα επιθυμούσα να ήταν λίγο πιο συγκεκριμένη η έκθεση σε ό,τι αφορά την παράγραφο 34 συγκεκριμένα Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, παράσχει αξιολογήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ε, σχεδίων υποδομών. Δεν αναφέρουμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εκπλήρωσε το καθήκον της για την παροχή αμερόληπτων αντικειμενικών ε, περιβαλλοντικών μελετών για τον αγωγό Nord Stream. Και ζητούμε όλα τα κράτη της Βαλτικής να συνυπογράψουν, προσυπογράψουν ε, την ε, σύμβαση ΕΣΠΟ. Νομίζω ότι και η Ρωσία όμως πρέπει να προσυπογράψει αυτή την σύμβαση γιατί έτσι θα εκπληρωθεί ο στόχος που έχουμε θέσει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μετσόνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υποστήριξα αυτή την πρόταση ψηφίσματος. Είναι σημαντική η πρωτοβουλία προωθείται από χώρες της Βαλτικής και τώρα υπάρχει αυτή η έννοια πια των μακροπεριφερειών. Είναι χρήσιμη η πρωτοβουλία πολιτικά και στρατηγικά. Υπάρχουν ουσιαστικά θέματα εδώ που είναι μέρος της επιχειρησιακής στρατηγικής της περιοχής και πάνω απ' όλα είναι σημαντικό το γεγονό ότι τώρα υπάρχει μια προοπτική, γιατί με αυτή την πρωτοβουλία δημιουργούμε τα θεμέλια για την ε, δημιουργία άλλων μακροπεριφερειών, μακροπρόθεσμα. Θα είναι αυτή η εμπειρία ένα πιλωτικό πρόγραμμα στην πραγματικότητα ως βάση για την έναρξη και το τρέξιμο και άλλων προγραμμάτων στα πλαίσια του, προγρα... του Ταμείου Συνοχής. Είναι σημαντικό και θα πρέπει η Κομισιό να δώσει μεγαλύτερη σημασία στην οικονομική προοικοδότηση αυτού του προγράμματος. Βέβαια υπάρχουν επιφυλάξει όταν πρόκειται για προσθήκη κονδυλίων, αλλά από την άλλη, χωρίς χρηματοδότηση, αυτά τα μεγάλα προγράμματα για τις μακροπεριφέρειες δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρξει κανονισμός για την οικονομική χρηματοδότηση αυτής τη πολιτική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μαντσόνη. Το λόγο έχει η ε, κυρία λένε. είναι εδώ. Ευχαριστώ. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή και χαίρομαι που εγκρίθηκε τελικά. Η έκθεση αυτή μιλάει για τη στρατηγική της Βαλτικής θάλασσας και παρατρύνει τα κράτη-μέλη να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους ανάλογα με και με την εδαφική ανάπτυξη. Γίνεται λόγος για πολλές δραστηριότητες. Μία από αυτές είναι η οικολογική δραστηριότητα. Και χαίρομαι που εγκρίθηκαν οι τροπολογίες μου. για την αξιολόγηση των ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις ε, υποδομές και στα ενεργειακά προγράμματα. Πιστεύω ότι με βάση τη στρατηγική αυτή για τη Βαλτική θάλασσα θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και με τις τρίτες χώρες. Και χαίρομαι που με την ενδιάμεση αναθεώρηση αυτής της ε, στρατηγικής θα έχουμε βαδίσει πολύ δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Περνάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Κράτσα το λόγο έχει πρώτη η κυρία Βάιντερε. Κυρία Πρόεδρε, ήθελα να μιλήσω κι εγώ για τη Βαλτική και τη στρατηγική για τη Βαλτική. Μπορώ να έχω το λόγο επ' αυτού. Κυρία Κουάντρας, μπορώ και εγώ να πω κάτι για τη στρατηγική της Βαλτικής, γιατί για εκείνο ζήτησα το λόγο. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Μιλήστε για τη Βαλτική. Για τη στρατηγική για τη Βαλτική θάλασσα, η περιοχή της Βαλτικής ε, ε, κρύβει πολλές δυνατότητες ανάπτυξης και αυτή η στρατηγική έχει δεχτεί οι υποσχέσεις για χρηματοδότηση. Θέλουμε μια δομή που θα συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής. Συντονισμένα προγράμματα εργασίας για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, για τις καινοτομίες στην έρευνα. Και έχουμε προβλέψει και μια ενιαία πολιτική έβραση τεχνιών για την περιοχή της Βαλτικής. Θέλουμε συνεργασία καλύτερη μεταξύ των επιστημόνων, να την προωθήσουμε και η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται πολύ από αυτή τη στρατηγική. Το πρόγραμμα της Βαλτικής έχει μπει στον πάγο και θα πρέπει να αναθερμανθεί και να προχωρήσει. Τα προγράμματα για τις καινοτομίες και των υποδομών θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Γι' αυτό υποστήριξα και το, την έκθεση. Τώρα θέλω να κάνω μια δήλωση για την έκθεση της κυρίας Κράτσα. Παρακαλώ, λέει ο πρόεδρος. Α, θα μιλήσετε για την έκθεση της κυρίας Κράτσα. Πολύ ωραία. Ακόμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην περιφερειακή πολιτική. Η πολιτική συνοχής και ο στόχος 2 προβλέπει βοήθεια στις περιφέρειες με υψηλή ανεργία και μετανάστευση. 54,7 εκατομμύρια δόθηκαν, αλλά ακόμα οι διαφορές είναι μεγάλες. Οι πιο φτωχές περιφέρειες ήταν αυτές που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση. Χρειάζεται βοήθεια, η βοήθεια πρέπει να δοθεί κατά προτεραιότητα. Πρέπει να παραμείνει αυτό προτεραιότητα. Θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά δίκαιος. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να δώσουμε υποστήριξη και στην περιφερειακή πολιτική και ιδιαίτερα να στηρίξουμε τις περιφέρειες όπου ε, οι μέσοι δείκτες είναι κάτω από τους ε, μέσους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά. Πρέπει να δράσουμε με τρόπο τέτοιο ώστε να δώσουμε πρακτική βοήθεια και να υποστηρίξουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα αυτοί που εργάζονται με οικονομικό και καινοτόμο τρόπο. Αυτοί χρήζουν μεγάλη ε, υποστήριξης. Μας εντυπωσιάσατε με τη γνώση των προηγουμένως με τις γνώσεις των αρχαίων Ελλήνων και της αρχαιολογικής τραγωδίας. Ποιες είναι οι πιο εύπορες ε, οι πλούσιες χώρες Ευρώπης ή με τους πλουσιότερους πολίτες. Κοίταξα τα έγγραφα του ΩΣΑ και το 2008 που είναι το τελευταίο έτος για το οποίο έχουμε στοιχεία. Οι χώρες με τους πλουσιότερους πολίτες είναι οι, τα μέλη της συμφωνία ε, Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου, άσχετα με τη χρηματοπιστωτική κρίση που έπληξε δυσανάλογα την Ισλανδία και την Ελβετία, το κατακεφαλήν εισόδημα στις χώρες ΕΖΕΣ είναι 214% ψηλότερο από τη... των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δύο φορές πιο πλούσιοι από εμά ε, οι πολίτες χώρες ΕΖΕΣ από τους πολίτες των Ευρωπαίων πολιτών. Άρα κάπου το πρόβλημα βρίσκεται στη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι μεν ε, μέσα σε πολλές ε, συμφωνίες, σε κοινέ πολιτικές, αλλά δεν είναι στην ε, κοινή γεωργική πολιτική, την αλληλευτική, τα ενεργειακά τους θέματα τα λύνουν μόνο τους και τα ανθρώπινα δικαιώματα επίσης έχουν δικές τους συμφωνίες. Δεν θα μπορούσε το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει κάτι αντίστοιχα καλό με αυτό που επέτυχαν 7 εκατομμύρια Ελβετοί και 4 εκατομμύρια Νορβηγοί. Γιατί θα μπορούσαμε κι εμείς να έχουμε αντίστοιχες επιδόσεις και να διαχειριζόμαστε τα δικά μας προς το δικό μας συμφέρον και όφελος όπως κάνουν και άλλοι. Thank ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όποτε μιλούμε για την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, είναι σημαντικό να ανατρέχουμε προς τα πίσω και να διδασκόμαστε κάποια πράγματα. Δηλαδή, τι έφταιγε, η μη κατάλληλη νομοθεσία της ΕΠΑ οδήγησε στις τράπεζες να δανείζουν επισφαλείς ε, ε, χρεώστες και να μην μπορούν να αποπληρωθούν τα δάνεια αυτά. Αυτά τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε όλοι. Ποιες είναι, λοιπόν, ποια είναι τώρα τα αποτελέσματα από τις χώρες που τυπώνουν χρήμα, αλλά σαν να μην έχει καμία αξία. Ο μόνος όμως οικονομολόγος που προέβλεψε την κρίση είχε πει ότι το χρήμα έχει αξία. Και με το φθηνό ε, χρήμα γίνονται επενδύσεις κακές ε, που δημιουργούν ε, την χρηματιστηριακή φούσκα που οδηγεί σε κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματο. Αυτό κάναμε και έτσι ξεκίνησε και το χρηματοπιστωτική κρίση. Ελπίζω να διδαχθούμε από τα λάθη παρελθόντος. Ευχαριστούμε πολύ. Έκθεση τώρα Καντσιάν και δίνω το λόγο στον κύριο Μικολάτσικα. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, η έκθεση Κάντσιαν για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν δεν καλύπτει άτομα με ειδικέ ανάγκες που ακόμα υφίστανται διακρίσεις. Η ίση πρόσβαση στις μεταφορές είναι προϋπόθεση για την ισότητα των ευκαιριών. Τύφλοι, άνθρωποι με προβλήματα όρασης ακόμα έχουν προβλήματα με τα λεωφορεία και τα πούλμαν. Εγώ χαιρετίζω τις τροπολογίες που ενισχύουν τα δικαιώματα ατόμων με ειδικές ανάγκες και ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα. Ιδιαίτερα καλωσορίζω τις διατάξεις για ειδική κατάρτιση ε, του προσωπικού που είναι στους σταθμούς λεωφορείων και πούλμαν για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Ευχαριστούμε κύριε Μικοάσικ. Το λόγο και κυρία Ρόιτοβα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έδειξε και σε, ότι σε αντίθεση με το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αντιληφθεί σωστά τις προτεραιότητες για τα δικαιώματα των επιβατών που δικινούνται με λεωφορεία και πούλμαν. Χάρη στην έκθεση αυτή λαμβάνουμε υπόψη και τα δικαιώματα των επιβατών με ειδικέ ανάγκες ε, και με ε, αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα. Πρόκειται για το άρθρο 11. Τώρα θα πρέπει υπάρχει των υπηρεσιών να εξασφαλίζουν δωρεάν παροχή βοήθειας καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, όπως και στις αεροπορικές μεταφορές. Έτσι θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων με αναπηρίες. Πρόκειται για ε, μία πρόκληση που στείλαμε προς το Συμβούλιο και ελπίζω να μην αποδυναμωθεί η θέση του Κοινοβουλίου στη δεύτερη ανάγνωση. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ. Εγώ τάχθηκα υπέρ της τροπολογίας 15 γιατί είμαι υπέρ της ε, χρονικά περιορισμένης εξαίρεσης για τις ε, χώρες τοπικές, αστικές και περαστικές μεταφορές, γιατί μερικές από τις απαιτήσει θα δημιουργήσουν τεράστιο κόστος για τις ε, εταιρείες μεταφοράς, ιδιαίτερα όταν είναι μικρομεσαίες και είναι υπερβολικό το άχθος. Κάτι που θα οδηγήσει στην εξαφάνισή τους από ορισμένε ε, αγορές και θα αποβεί βάρος των πελατών γιατί θα χάσουν κάποιες τοπικές μεταφορές, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Γιατί εντάξει να μιλούμε για αστικέ και περαστικέ μεταφορές, αλλά στις τοπικές μεταφορές, στην Ήπεθρο, θα δημιουργηθεί κίνδυνο αν είμαστε τόσο απαιτητικοί στι προϋποθέσεις. Θα οδηγήσουμε στην εξαφάνιση πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εξασφαλίζουν αυτέ τι τοπικέ μεταφορέ. Είπαμε να μην υπερφορτώνουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει με υπερβολικό άκθο και νομίζω ότι δεδομένης κατάστασης μια λογική συμβαστική λύση θα ήταν μια προσωρινή εξαίρεση για τις περιπτώσεις αυτές. Παίρνουμε τώρα στην έκθεση Στέρξ. Το λόγο έχει ο κύριος Λαβία. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης για το την υποβολή δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλο ή απόπλου από τους λιμένες γιατί έτσι θα διευκολυνθούν οι παράκτιες μεταφορές. Τώρα υπάρχει πολύ γραφειοκρατία περιπλοκή και προστίθεται και η έλλειψη εναρμόνισης στο πειθαρχικό τομέα και το πώς θα εφαρμόζεται η, από τα κράτη-μέλη του 2002 η οδηγία. Χρειάζεται λοιπόν μια οδηγία πολύ λεπτομερής που θα μειώνει στο ελάχιστο τις παρερμηνίες. Ε, βέβαια θα πρέπει να απλοποιηθούν και οι διοικητικέ διαδικασίες με νέα νομοθεσία που θα, ε, ώστε να λαμβάνονται υπόψη ε, τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφοριών. Είναι καλό να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών εδώ. Περνάμε στην έκθεση Gross. έχει το Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο τομέας των μεταφορών είναι από τους τομείς όπου, που επηρεάζεται από πολλά θέματα. Κύρια σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την υγεία, την ανταγωνιστικότητα, της ενιαίας αγοράς, την ε, οδική ασφάλεια κλπ. Ε, ενίσχυση διαφορετικών οργανισμών για τις διάφορες μεταφορές, τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, τις εκπομπές. Γι' αυτό λοιπόν είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει στρατηγική για τις μεταφορές που θα διασφαλίζει την βιωσιμότητα, τη σταθερότητα μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό, δημοσιονομικό πλαίσιο. Γι' αυτό είμαι υπέρ της έκθεσης Γκρός και θέλω να τον, να τον συγχαρώ για την εργασία του. Ευχαριστούμε. Κυρία Μουσκαρντίνη τώρα έχει το λόγο. Δεν βλέπω να είναι στην αίθουσα. Κύριο Στάκουλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε για την αηφόρο ανάπτυξη στις μεταφορές. Πρέπει να το διασφαλίσουμε αυτό αφού θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι οι βλάβες λόγω των μεταφορών, οι ρήποι θα μειώνονται συνεχώς στο μέλλον. Γιατί οι μεταφορές μπορεί να είναι ένα μικρό κομμάτι στην οικονομία μας, αλλά για αηφόρο μέλλον χρειάζεται και ε, βιώσιμες μεταφορές θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες παντού στην Ευρώπη, γιατί εδώ εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα ακόμη. Είναι διαφορετικές οι διατάξεις ε, στις διάφορες περιφέρειες και κράτη-μέλη της Ένωσης ε, και εδώ χρειάζεται εναρμόνιση. Οι ίδιοι κανόνες να ισχύουν παντού. Είναι επίσης ε, σημαντικό να επενδύσουμε στις τεχνολογίες, στις ε, καινοτομίες, στην ανάπτυξη ε, και για το μέλλον των μεταφορών σημαντικό αυτό. Περνούμε τώρα στην έκθεση Τουργκάιθ. Το λόγο ο κύριος Μαστέλα. Ευχαριστώ. Η θέση ισχύει της συνθήκης της Λισαβόνας επανεπιβίωσε το δικαίωμα της αναφοράς που είναι θεμελιώδη στοιχείο της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Αναφίβολα το δικαίωμα της αναφοράς είναι το εργαλείο που εξασφαλίζει στου πολίτες να καταθέσουν στους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες τις ανησυχίες σε σχέση με τις διάφορες πολιτικές ή νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς επηρεάζει την καθημερινότητά τους. Υπάρχει όλο και αυξανόμενος αριθμός αναφορών για το περιβάλλον, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δικαιοσύνη, την ενιαία αγορά, την ανάπτυξη κτλ. Όπως είδαμε και από τις ε, προηγούμενες εκθέσεις, μπορούμε να περιμένουμε μια καλύτερη θεσμική, διαθεσμική συνεργασία και επικοινωνία σε ό,τι αφορά το μηχανισμό καταγγελίας των Ευρωπαίων πολιτών. Χρειαζόμαστε μια ενιαία θηρίδα ώστε να μπορεί σε ένα σημείο να αποτείνεται ο Ευρωπαίος πολίτη και να βρίσκει λύση στο πρόβλημά του καταγγέλλοντα μια παραβίαση δικαιώματο. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πιο διαδραστικό, ε, μια πιο διαδραστική ιστοσελίδα που να ενημερώνει τους πολίτες πριν ε, αποφανθούν ποιο είναι ο κατάλληλο μηχανισμό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Κύριε Σακάλα, για αυτή... κύριε Σον Κέλλη, για αυτή την έκθεση, μια στιγμή προηγείται κυρία Βάιντερε και μετά εσείς κύριε Κέλλη. Κυρία Βάιντερε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Μεταφορών ε, πήραν 1924 αναφορές και το 46% μόνο έγινε, κρίθηκε παραδεκτό και δόθηκε συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν έχουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με το πώς απευθείας μπορούν να προσεγγίσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα προέτεινα η ιστοσελίδα της Επιτροπής Μεταφορ... Ε, Αναφορών να βελτιωθεί γιατί Πολλοί άκουσαν ότι μπορούν να ε, αξιοποιήσουν, για παράδειγμα, το σύστημα Solvit Online. Πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες και ιδιαίτερα και αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Η Επιτροπή Αναφορών είναι ο πιο γρήγορος δρόμος για να απευθυνθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι πολίτες και νομίζω ότι η δουλειά αυτή θα πρέπει να γίνει με ακόμα περισσότερη αίσθηση ευθύνη. Ευχαριστώ, γι' αυτό υπερψήφισα. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ, είστε πολύ ευγενικό. Η Επιτροπή Αναφορών είναι από τις επιτυχίες της Ένωσης και εγώ και άλλα μέλη το είδαμε αυτό γιατί παρέχονται συμβουλές, υποστήριξη και ένα ευήκον ους προς ανθρώπους που αντιμετώπισαν γραφειοκρατίες στη χώρα τους και απογοήτευση και εκνευρισμό πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα για να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας, να επικοινωνούμε τα μηνύματα καλύτερα στους πολίτες, να επιταχύνουμε τη διαδικασία και τρίτον, τα κράτη-μέλη πρέπει να αναγκαστούν να απαντούν σε ερωτήματα πιο γρήγορα από ό,τι κάνουν τώρα, γιατί ε, ταλαιπωρούν τη διαδικασία με τις καθυστερήσεις, τις απαντήσεις και αυτό δεν δημιουργεί ικανοποιητική κατάσταση. Αλλά αυτό είναι καλή εξέλιξη και ε, χαίρομαι την Επιτροπή που έτεινε βίκον ούς ανθρώπους που το, χρειαζόταν, το χρειάζονταν. Ευχαριστώ κύριε Γκέλη. Κύριε Γκέλη, την άλλη φορά μην ξεχάσετε από πριν αρχίσω με τις επεξηγήσεις ψήφου να μπείτε στον κατάλογο γιατί δεν είσαστε στον κατάλογο, γι' αυτό δεν σας έδωσα το λόγο. Εντάξει, εντάξει, πήρα το μάθημά μου. Περνάμε τώρα στην έκθεση του Ρουνέν η κυρία Ροντσούλη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η οικονομική κρίση έπληξε τους ε, Ευρωπαίους νέους ε, με πολύ πιο έντονο τρόπο δυσκολεύοντας ε, τις προοπτικές τους. Ε, ένα μεγάλο ποσοστό των νέων από 18-25 ετών, ε, ένα στρατός 5,5 εκατομμυρίων νέων δηλαδή, δεν μπορούν πλέον να βρουν θέση απασχόλησης. Οι δημογραφικές και οικονομικές προοπτικές για την επόμενη πενταετία δυστυχώς προβλέπουν τη δημιουργία 8 εκατομμυρίων θέσεων εργασία στην Ευρώπη που στις περισσότερες περιπτώσεις θα απαιτούν πολλά προσόντα. Επομένω, αυτή είναι η πρόκληση για του νέου μα και αυτή είναι και η μόνη επένδυση που θα εγγυηθεί ε, ένα μέλλον για αυτού του νέου. Αρκεί να δει κανεί ε, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την ε, επονίδιστη θα έλεγα μετάλλευση που υφίστανται ορισμένοι νέοι. Στόχο είναι να, η ανάκαμψη τη απασχόληση, Νομίζω όμω ότι θα πρέπει το επίκεντρο να είναι οι νέοι, οι ανάγκες τους και οι προσδοκίε του. Ευχαριστούμε κύριε Ραντσούλη. Το λόγο κύριο Στάκουλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ζωτική σημασία να διευκολύνουμε τους νέους στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Ήταν πολύ καλή έκθεση του Ρούνεν από την άποψη αυτή και χαίρομαι που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται να αλλάξει η νοοτροπία μας, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στα κράτη-μέλη. Γνωρίζουμε ότι η ανεργία της νεολαίας έχει ξεφύγει από τον έλεγχό μας. Μιλούμε για αστρονομικά ποσοστά, 20%. Δεν είναι σωστός αυτό, σωστή αυτή η εξέλιξη για το μέλλον. Χρειαζόμαστε κάποια μέτρα χρήσιμα στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Δεν χρειαζόμαστε ωραία λόγια μόνο και αγαθές προθέσεις. Χρειαζόμαστε έργα, γιατί οι νέοι μας μένουν άνεργοι οι νέοι μας δεν έχουν την πείρα που χρειάζονται για να προσληφθούν. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποιους δρόμους, κάποιες δυνατότητες να φέρουμε τους νέους στην αγορά εργασίας και να έχουμε μια πιο αηφόρο αγορά εργασίας στο μέλλον. Ελπίζω ότι δεν θα αρχιοθετηθεί η έκθεση αυτή απλώς, αλλά πραγματικά θα οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης των νέων. Η κυρία Ουρκουλέιτε. Ευχαριστώ κυρία, κύριε Πρόεδρε. Ε, η ανεργία των νέων είναι πολύ πιεστικό πρόβλημα σήμερα γιατί 20% ανθρώπων στην ηλικία μου δεν έχουν δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ψήφισα υπέρ της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί νομίζω ότι αποστέλνουμε ένα ακόμη σημαντικό μήνυμα και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη για την κατάσταση τη, στη, της ανεργίας των νέων. Συμφωνώ με την έκθεση ότι προγράμματα όπως το ΕΡΑΣΜΟΥΣ για τους νέους επιχειρηματίες πρέπει να τύχουν στήριξης μεγαλύτερης. Είναι σημαντικό να τονίσουμε την σημασία της άτυπης εκπαίδευσης, κατάρτισης των νέων. Επίσης πρέπει να μας απασχολήσει και η στρατηγική 2020 γιατί η ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας θα πραγματοποιηθεί και μέσα από πράσινες θέσεις εργασίας. Η Λιθουανία έχει δημιουργήσει κάποιες ευνοϊκές συνθήκες ήδη για τις επιχειρήσεις που απασχολούν για πρώτη φορά τους νέους, που, νέους ερχόμενους δηλαδή στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε στην έκθεση Γκρουνή. Κυρία Ρούντσουλη, το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. πιο ευέλικτες μορφές εργασίας γενικά δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων. Οπότε αυτές οι επισφαλείς θέσεις εργασίας πρέπει να αντιμετωπιστούν από εμάς στο Κοινοβούλιο για να έχουμε ε, τη δυνατότητα να προσφέρουμε μεγαλύτερη ασφάλεια σε όλους τους εργαζομένους αυτή η έκθεση θα μας βοηθήσει η δυνατότητα εξέβρεσης εργασίας με καλές μελλοντικέ προοπτικές. Αυτό είναι ο σημαντικότερος στόχος, ώστε η ευρωπαϊκή ε, οικονομία να ανακάμψει. Ελπίζω όλα τα κράτη-μέλη να επενδύσουν περισσότερους πόρους ε, στο θέμα αυτό για να πούμε ναι στην Ευρώπη της γνώσης και της απασχόλησης και όχι στην ευρωπαϊκή επισφάλεια. Περνάμε στη τελευταία έκθεση, την έκθεση του κ. Φερνάνδη δηλαδή. Ο κύριος Πυρίλο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η σημερινή ψηφοφορία από τις εκθέσεις Φερνάντες ήμουν σκιώδης εισηγητή ε, για την ε, ομάδα μου συγκεκριμένα ε, δείχνει με σαφή τρόπο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει από την Εκτελεστική Επιτροπή να καταθέσει ειδική οδηγία για τα βιολογικά απόβλια, για τη διαχείριση των βιοαπικοδομήσιμων ε, αποβλήτων και για την διαφοροποιημένη συλλογή, κάτι που θα είναι υποχρεωτικό με την καλή διαχείριση τα με απόβλητα μπορούν να γίνουν μια ε, σημαντική πηγή παραγωγή ε, βιοαερίου συγκεκριμένα, μια ανανόσιμη πηγή ενέργεια πολύ σημαντική που μπορεί να δημιουργήσει, να μετα... Ε, σε βιομεθάνιο παραδείγματο χάρη και ακόμη και να παραγάγει ηλεκτρική ενέργεια. Υπήρξαν ιδιαίτεροι δισταγμοί από πλευράς Επιτροπής για την εκπόνηση οδηγίας, αλλά μαζί με άλλους συναδέλφους στείλαμε ε, στην Επίτροπο, την αρμόδια, τον στον αρμόδιο Επίτροπο μάλλον, τον κύριο Ποτότσινικ, τις προτάσεις μας ελπίζοντας ότι θα έχουμε το συντομότερο δυνατόν τις προτάσεις του. Κυρία Μουρκουνάη, την τελευταία ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα βιολογικά απόβλητα είναι ζήτημα για όλους τους πολίτες της Λιθουανίας γιατί η κατάσταση της διαχείρισης λιμάτων και αποβλήτων διαφέρει ε, στα κράτη-μέλη. Μερικοί ε, το 10% του, των αποβλήτων αυτών τα αφήνουν στις χωματερές ενώ άλλοι έχουν υψηλότερο ποσοστό. Θέλουμε να μειώσουμε το, τον όγκο των αποβλήτων και επιπλέον να εμφυσίσουμε την ε, νοοτροπία της ανακύκλωσης όλο και περισσότερο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να μελετήσουμε όλες τις ε, συνθήκες ε, και τις επιπτώσεις για να αποφύγουμε την επιδείνωση της κατάστασης αυτής. Θα πρέπει να δούμε επίσης τι είδους βιολογικά απόβλητα θεωρούνται λίπασμα Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ρόιτοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία που μου δώσατε να κάνω την επεξήγηση ψήφου ό,τι αφορά την πράσινη βίβλο για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων. Συμφωνώ με το γενικό πλαίσιο. Γιατί πριν την ε, κατάρτιση μιας νομοθετικής πρότασης, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει πρώτα να ασχοληθεί με το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων και την κατάσταση ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει πιο ε, διεξοδικά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της ε, καλλιέργειας ε, των τροφίμων, των ε, προϊόντων για βιοκαύσιμα. Επίσης το θέμα της αποθήκευσης και της διαχείρισης με απασχολεί ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε για το μεσημέρι.